Eh, vabbè. Vai, ogni giorno la sua pena. Dear colleagues, good evening. I would like to start... Καλησπέρα συνάδελφοι. Uh, with, uh, adopting the... Έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Ξεκινάμε. Εγκρίνεται, ευχαριστώ. Δεν έχω ανακοινώσεις, τίποτα. Πάμε λοιπόν. στο σημείο υπαρίθ 4 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση Ιάκωπ Φον Βάιτσακα επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κρατικά ομόλογα και τίτλους των τραπεζών. Πολύ σημαντική πρόταση. Έγινε η παρουσίαση της εκθέσεως, υπευλήθησαν οι τροπολογίες, βρισκόμαστε στη φάση συζητήσεων των τροπολογιών. 197 τροπολογίες έχουμε. Ε, ε, να ζητήσω τον Ιάκοπ Φον Βαϊτσέκα να πάρει το λόγο και να τον συγχαρώ για τη μελλοντική του θέση επί τη ευκαιρία σημαντικότατη. Είμαι θα υπερήφανη πλευρά οίκων για την επιφανή θέση που θα κατέχει από τούδε και στο εξή ένα μέλος της οίκων. Τώρα είσαστε εδώ, υπό την παρούσα σας ιδιότητα, του Ευρωβουλευτού και του Συγητού. Γιάκοπ λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Πράγματι, πράγματι συζητούμε ένα πρόβλημα εδώ και τις τροπολογίες αυτού. Είναι σκληρό πρόβλημα. Πάει στην καρδιά του προβλήματος για το πρόβλημα των ομολόγων, των τραπεζών και των κρατικών ομολόγων. Γι' αυτό είχαμε και 197 τροπολογίες. Είχαμε και διάφορες τροπολογίες για απορρίψει θυμάτων του κειμένου. Είναι γιατί είναι το σκληρό το πρόβλημα. Κάποιες τροπολογίες για απορρίψει προχώταν εξ αριστερών, άλλες εκ δεξιών. Και αυτοί με τους οποίους συνομίλησα, ενώ απορρίπτουν, ε, απορρίπτουν την πρόταση, δεν έχουν δώσει κάποιες πιστικές εναλλακτικέ για το πρόβλημα αυτό. Um, um, για το πρόβλημα αυτό των τραπεζών. Άρα μέλη, πέρα από αυτό, έχουν υποβάλει πάνω από 130 τροπολογίες για να συμβάλλουν επικοδομητικά, ούτως ώστε να βελτιωθεί η έκθεση. Με τα χαράς σας αναφέρω ότι έχουμε μεγάλο αριθμό ενδιαφερουσών τροπολογιών που εκτιμώ και σε πολλούς τομείς θα πρέπει να είναι εύκολη μια συνένεση μεταξύ αυτών που υπέβαλαν κάποιες τροπολογίες κάποια τμήματα. Θα αναφέρω κάποιους τομείς όπου δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα συνένεσης. Πιστοποίηση και εποπτεία είναι ένας τομέας χρειάζεται μια στάθμιση. Η εξουσία της ΕΣΜΑ από πλευράς επιστοποίησης και εποπτείας. Κάτι που ξεπερνά τα προτινόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα της οριμότητας ε, και των διαφόρων στοιχείων του, του μη χρησιμοποιημένων στοιχείων ενεργητικού. Και είναι ένας τομέας όπου δεν έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λύσεις και έχουμε και το θέμα της αναδιάθρωσης του χρέους, που δεν έχει καν πρόβλημα. Σε κάποια θέματα μπορούμε καλές λύσεις. Μετά να δούμε ποια είναι η όλη διάθρωση του θέματος, ο αριθμός των δόσεων των τμήματων, Λοιπόν, ε, να έχουμε τρία επίπεδα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλοι θέλουν δύο επίπεδα, αλλά δεν είναι μόνο ο αριθμός των επιπέδων, αλλά και το μέγεθος αυτών, των τμήματων. Πολλές ιδέες υπάρχουν. Από άκαμπτες προϋποθέσεις διαχωρισμού, μέχρι την ιδέα ότι δεν πρέπει να καθοριστεί τίποτα και όλα να αφαιθούν στη διάκριση της αγοράς. Μεγάλη ποικιλομορφία προτάσεων. Εγώ είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο ότι με τις υποβληθεί τροπολογίε θα βρούμε λύση. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση επί του χαρτοφυλακίου του SBBS. Θα μπορούσε και αυτό να αφαιθεί στις αγορές. Άλλη ιδέα ήταν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αναλογία με την κλίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά με το εκκρεμόν χρέος. Αυτό ίσως να δημιουργήσει απορίες κάπου. Είναι μια πρόταση όμως που υφίσταται. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου και σχέση με αυτό πώς αποφασίζουμε και βάσει πριν κριτηρίων πότε να υπάρχει απόκληση από οποιαδήποτε κλίδα χαρτοφυλακίου επιλέγεται. Σε περίοδους κρίσεων, απώλεια πρόσβαση στην αγορά, ένα θέμα, άλλο θέμα, αρνητικός αντίκτυπος στη ρευστότητα της αγοράς, για το εθνικό τμήμα του χρέους εκτός του SSB. Χρειάζονται τεχνικής φύσεως συζητήσεις θα ήταν χρήσιμες. Μπορεί να επιληθεί το θέμα όμως. Και ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που είναι πολιτικής φύσεως. Αν το SBBS θεωρηθεί χρήσιμο στοιχείο για αυτό το γκόμβο αυτό των ε, τραπεζών, σε ποιο βαθμό αυτό το δίπολο και πέρα από την δημιουργία βάσεως μέσω νομοθεσίας, με την δημιουργία του SBBS αν μπορεί να υπάρξει κρίση και αξιολόγηση πώς τα τμήματα του SBBS ε, να βάλουν υπόψη στο ισοζύγιο των τραπεζών. Εγώ ήθελα να παραμείνω ανοιχτό στο θέμα. Δεν θα ήθελα οι τράπεζε όμως να χρησιμοποιήσουν το κατώτερο επίπεδο, το ελεγχόμενο τμήμα του SBBS, για να μειώσουν το ισοζύγιο του, αναλαμβάνοντα μεγαλύτερο χρέος να φάτε κατοικά ομόλογα από ό,τι μέχρι τώρα. Γι' αυτό προσπάθησα να διατηρήσω την καθιστική ατάξη και να μην ενθαρρύνω πιο ρηψοκίνδυνη συμπεριφορά. Δηλαδή ότι το κρατικό χρέος με το θεωρήμα με την επιχείρημα ότι το κρατικό χρέος οι τράπεζες το αντιμετωπίζουν στα πλαίσια μελλοντική νομοθεσίας. Άλλοι λένε ότι το αντιμετωπίσουμε τώρα, οριστικά και τελειωτικά. Περιορίζοντα τη δυνατότητα που έχουν οι τράπεζε να έχουν SBBS, και να το εντάσσουν στο ανώτερο επίπεδο τώρα. Είναι θέμα κρίσης. Εμείς τι θεωρούμε ότι πρέπει να κάνει αυτή η νομοθεσία. Και αργότερα τι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει. Στα πλαίσια ενό μεγαλύτερου παζαρέματος τι θα πρέπει να αποφασιστεί επί του κρατικού χρέους. Η ρυθμιστική προσέγγιση του SBBS θα είναι αντικείμενο πολιτικών κολλημάτων. Εγώ ίδιος δεν θα δεχόμουν μια λύση κατά την οποία οι τράπεζες θα μπορούν να έχουν πιο επικίνδυνη συμπεριφορά σαν αφορά τα κρατικά ομόλογα από ό,τι τώρα. Αλλά εγώ θα ήμουν στεναρά υπέρ προσεγγίσεως δύο βημάτων. Θα πούμε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος των κρατικών ομολόγων στις τράπεζες δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στο SBBS, δεν είναι αρκετά ευρύ. Οπότε το SBBS και ο κίνδυνος από τα κρατικά ομόλογα θα αντιμετωπιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Σταματά εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το λέω έχουν οι σκιώδεις εισηγητές. Υπάρχει κάποιος από το ΕΛΚ. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποια διαφάνεια, οπότε δεν ξέρω γιατί κατεβαίνει η οθόνη, εκτός αν θέλουμε σκιά για αυτούς τους σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελε λοιπόν κάποιος το λόγο εκ μέρους του κυρίου, του κυρίου Σέλο από το ΕΛΚ. Έχω μία δήλωση του κυρίου Λούκε, εξ ονόματος της ομάδας ECR. Μου ζήτησε να την διαβάσω. στα αγγλικά. Μπορώ να το κάνω αν χρειαστεί. Ε. Oh, of course I'm not. Uh, Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Πιστέψτε με, δεν συμφωνώ με αυτό που θα διαβάσω, μπορώ όμως ε, να διαβάσω το κείμενο του κυρίου Λούκε για να είμαστε δίκαιοι. Θα συνοψίσω λοιπόν, διότι το κείμενο είναι πολύ μεγάλο. Ο εισηγητής ε, στην ουσία έχει αρκετές αμφιβολίες, όχι με συγχωρείτε, ο σκιώδης εισηγητής έχει αρκετές αμφιβολίες, διότι θεωρεί ότι είναι ένα πάρα πολύ προβληματικό ζήτημα και θα ήθελε λοιπόν ιδανική ε, ανοχή για, την, για το κατώτερο τμήμα. Ο, ο κύριος Λούκε φοβάται ότι το συνολικό ομόλογο θα λάβει μηδενική εξασφάλιση κινδύνου σε αυτήν την περίπτωση. Και έτσι θα διευρυνθούν τα προνόμια αντί να μειωθούν. Γι' αυτό λοιπόν η ομάδα ECR έχει αρκετές αμφιβολίες για τις ε, τροπολογίες αυτές. Ο, κύριος Λούκη θεωρεί πως ε, πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που επιθυμεί η ομάδα ECR και αυτό είναι σε γενικές γραμμές οι απόψεις του. Είναι πολύ σημαντικό να τι ακούσουμε για να γίνει συζήτηση. Βέβαια καλό θα ήταν να είναι εδώ και ο εισηγητή, αλλά νομίζω πως ε, μπορούμε τουλάχιστον να ακούσουμε την άποψή του. Αυτά λοιπόν ε, εξ ονόματος της ομάδας ECR και ο κύριος Καλβέ Σαμπόν, εξ ονόματος των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσω τη γλώσσα του Θερβάντες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, καταρχήν, και να πω ότι υπήρχαν τροπολογίες από τη δεξιά, από την αριστερά και από τους φιλελευθέρους που είμαστε και το μόνο μέλλον, εφικτό μέλλον. Έχουμε ένα επικοδομητικό όραμα για να προωθηθεί αυτό το πλαίσιο και ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι υποκατάστατο των ευρωομολόγων, όμως ε, είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο για να λάβουμε υπόψη τις διάφορες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Και για να μην ε, ε, δηλητριάζουμε τη σχέση μεταξύ τραπεζών και εθνικού χρέους. Φυσικά, Υπάρχουν ε, πολλές τροπολογίες που δεν μπορούμε να δεχτούμε και ε, μερικές επικοδομητικές. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να δεχτούμε πολλά από τα θέματα του κυρίου Βάισάκερ μέσα στα πλαίσια των διαφόρων κατηγοριών. Εάν αυτά τα στοιχεία ενεργητικού κινηθούν προς το κοινό γενικότερα και τις ε, επενδύσεις ε, μικρής ε, εμβέλειας, τότε θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα μερίδια της αγοράς και πώς θα κατανεμηθούν μέσα στα πλαίσια των επενδυτών αγοράς. Αυτό είναι ένα θέμα που θέτουμε επιτάπητος. Αυτό το μέσο ε, υπάρχει. Αν θέλετε το διαχωρίζουμε σε δύο, τρία ή τέσσερα μέρη. Εμείς θεωρούμε και υποστηρίζουμε ότι η αρχή έκδοσης θα πρέπει να έχει λάβει ορισμένες ε, δεσμεύσεις. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι μέσα στα πλαίσια του τραπεζικού ή χρηματοπιστωτικού συστήματος, έτσι ώστε να υπάρχουν εγγυήσει. Πρόκειται για μία ανοιχτή συζήτηση. Αυτό που έχει σημασία είναι να ε, μπορέσουμε να επιβλέψουμε τις ε, εκδούσες αρχές και αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών. Γιατί μιλάμε για μία προστιθέμενη αξία που θα πρέπει να ε, προωθήσουμε. Γιατί άκουσα σήμερα ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών ε, δεν λαμβάνει υπόψη αυτό το πλαίσιο ελέγχου από πλευράς των ε, εκδίδουσών αρχών. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε σε, ένα, σε μια βάση στοιχείων ενεργητικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα ήθελα να προχωρήσω πιο μακριά. Και θα πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί έτσι ώστε τα θέματα αυτά να προωθηθούν ενεργά. Και αυτό και από πλευράς του κυρίου Βαϊσέκερ και των άλλων. Ευχαριστούμε. Θα μιλήσετε για τους πρασίνους, από τους πρασίνους. Καταρχήν, σε ε, μορφή προημίου, εάν κάποιος δεν θα μπορεί να έρθει εδώ, δεν θα πρέπει να σας δώσει ένα χαρτάκι να διαβάσετε και δεν ήξερα ότι ο πρόεδρος μπορεί να διαβάσει τα σημειώματα των βουλευτών σε σχέση με τον Ιακώμπ. Θα ήθελα να τον συγχαρώ για τη νέα του θέση και δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε αρχίσει τις ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβουλίο και χαίρομαι γιατί το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας θα έχει έναν άλλο φίλο Ευρωπαίο που είναι είδος ενεξαφανίσει Ελπίζω λοιπόν να μην ζήσει μεγάλες απογοητεύσεις. Τώρα θα, σα... σας διαβάσω το σημείωμα του κυρίου Όρτασον. Δεν μπορεί να είναι εδώ απόψε μαζί μας. Καθίσταται σαφές ότι δεν υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για αυτή την πρόταση και συμμεριζόμαστε αυτή τη στάση για διαφορετικούς λόγους από αυτούς που προέβαλαν οι άλλες, ομάδες. οι Δεν θεωρούμε ότι αυτοί οι τίτλοι ε, οι οποίοι ε, υποστηρίζονται από κρατικά ομόλογα μπορούν να υποστηρίξουν την Ευρωζώνη. Δεν είναι ένα μέσο που μπορεί να σταθεί από μόνο του, αλλά δεν πρόκειται και για ένα φιλόδοξο σχέδιο. Αντί να φτάσουμε σε δημοσιονομική ένωση και αμοιβεοποίηση των κινδύνων, το SBPS στην ουσία λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες ορισμένων μελών της Ευρωζώνης και όχι τη, πραγματική ανάγκη της Τραπεζικής Ένωσης. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξευρεθούν νέα τραπεζικά μέσα, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε για να τροποποιήσουμε αυτή την πρόταση, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας χωρίς να υπάρχουν αρνητικά αρνητικά σε σχέση με τη ρευστοποίηση των ε, ομόλογων των κρατικών ομολόγων. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχουν ε, τροπολογίες που είναι άκρος ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα οι 180 των σοσιαλιστών, και επίσης το ECR και οι φιλελεύθεροι ζητούν μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της ΕΣΜΑ και όχι των εθνικών αρχών. Είχαμε πολύ αρνητικές εμπειρίες στο παρελθόν από τις κρατικές αρχές και θεωρώ ότι ένα τέτοιο πανευρωπαϊκό προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται υπό τη ε, δικαιοδοσία της ΕΣΜΑ και αυτό αφορά και άλλα μερίδια της αγοράς, δηλαδή δευτερογενή μερίδια, τα οποία θα πρέπει να διέπονται από τις ίδιες αρχές. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, ρήτρε διασφάλισης για να μην έχουμε αρνητικές απόρριες στην αγορά κρατικών ομολόγων και για να μην υπάρχει έλλειψη ρευστότητας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να δούμε πώς προσδιορίζεται το χαρτοφυλάκιο. Θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένες σχέσεις μέσα στα πλαίσια της ε, κατανομής κεφαλαίου. Ε, Επίσης, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε χώρες από το χαρτοφυλάκιο αυτό. Υπάρχει αυτή η εναλλακτική, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα ε, στάθμισης του χαρτοφυλακίου. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε τα περισσότερα δυνατά στοιχεία μέσα στα πλαίσια των εκδόσεων ε, κρατικών τίτλων. Το SPS PBS είναι ένα νέο μέσο και δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι συνέπειες θα έχει. Θα πρέπει να υπάρχουν και ε, διορθωτικά μέτρα κατεπίγουσας ανάγκης εάν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στην αγορά ομολόγων κρατών μελών. Όπως βλέπετε στην τροπολογία μας, 181 στο άρθρο 90 θεωρούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θα πρέπει να ορίσει αυτή την αγορά χρεογράφων και σε περίπτωση κατεπίγουσας ανάγκης θα πρέπει να υπάρχουν προειδοποιήσεις και ενδιάμεσα μέσα έτσι ώστε να σταματήσουν να εκδίδονται κρατικά ομόλογα. Ε, εν πάση περιπτώσει θέλουμε να συνεργαστούμε επί του θέματος αυτού, αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία που χρήζουν βελτίωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Σίντοβαν, δεν σας είδα, είσαστε πίσω-πίσω. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μάλλον κάθομαι στην τελευταία σειρά και δεν φαίνομαι και αυτό είναι μια ένδειξη του ότι πρέπει να αλλάξουν οι πλειοψηφίες εδώ. Όμως, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον ε, Γιάκο, να τον συγχαρώ και για την έκθεση και για τη νέα του θέση στο Υπουργείο Οικονομικών. Νομίζω και ελπίζω να συνεργαστούμε καλά στο μέλλον. Η δική μου ομάδα κατέθεσε μια τροπολογία απόρριψης για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή νομίζω πως ε, τα SBPS δεν πρόκειται να εκπληρώσουν τον σκοπό τους, δεν πρόκειται να δώσουν ασφάλεια στους επενδυτές και μάλιστα θα συμβεί το αντίθετο. Θα κατευθυνθούν προ προς ε, πιο πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Έπειτα νομίζουμε πως, ε, τα, πως οι τίτλοι αυτοί δεν είναι οι κατάλληλοι για να αντιμετωπίσουν την ε, κρίση στην Ευρώπη. Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερες μακροοικονομικές ανισορροπίες και είναι επίσης μεγάλος ο κίνδυνος να είναι πολύ συνδε, ε, έντονα συνδεδεμένες με την ε, πολιτική λιτότητας. Ωστόσο, παρά την ε, τροπολογία απόρριψης, είμαι σε θέση να στηρίξω ορισμένα σημεία. Νομίζω πως η Γκουε θα μπορέσει να οδηγηθεί σε έναν συμβιβασμό για, σε ό,τι αφορά την αύξηση κατά 5% που, της, του κατώτερου τμήματος. Νομίζω πως ε, θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε αυτό το θέμα και είμαστε ε, διατεθειμένοι να συνεργαστούμε επικοδομητικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα νομίζω δεν έχουμε άλλους ομιλητές. Να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή για τα τελικά του σχόλια. Καλωσορίζοντας αντιπρόεδρο και επίτροπο, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπο του κ. Μοσκοβισή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους για τις επικοδομητικές τους συνεισφορές στη συζήτηση. Μπορώ να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι τελευταία φορά που θα ομιλώ εις αυτήν την Επιτροπή και τελευταία φορά που θα ομιλώ εις αυτό το Κοινοβούλιο. Κατέδειξε η συζήτηση ότι είναι υπέροχη αυτή η Επιτροπή μπορεί να συζητήσει και να διαπραγματεύεται πολύ δύσκολα χαρτοφυλάκια και να εξευρίσκει συμβιβασμού. Θα έχουμε μόνο μια συνεδρίαση σχεδόν αύριο εμεί. Ίσως δεν θα δω εγώ να ολοκληρώνεται η εξέταση του θέματος. Όμως η σύντομη αυτή συζήτηση έδειξε το πνεύμα που επικρατεί. Θα μου λείψει πολύ. Το λιγότερο μπορώ να πω είναι ότι ελπίζω ότι αν έρχεται στο Βερολίνο Κάποιοι από σας ζείτε και στο Βερολίνο. Χρησιμοποιήστε την ευκαιρία και ψάξτε να με βρείτε. Ελάτε να με βρείτε στη νέα μου θέση. Ένα ουσιαστικό σχόλιο. Δίκιο έχετε. Πράγματι. Μία σπιρίνη δεν μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο. Αλλά κάνει καλό μου στον πονοκέφαλο. Δεν πρέπει να κατηγορούμε την ασπιρίνη που δεν μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο αλλά να είμαστε ευχαριστημένοι που ασπιρίνη τουλάχιστον θεραπεύει τον πονοκέφαλο. Έχοντας αυτό υπόψη, μπορούμε να είμαστε πιο θετικοί. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι ισχυρό συστατικό για την αντιμετώπιση των ασθενειών της Ευρωζώνης. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει πανάκια με επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έξοχη δουλειά που κάνατε προσβλέπω σε μια εκ νέου συνάντησή μας ε, σε κάποιες άλλες ευκαιρίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Jacob. Ευχαριστώ, Γιάκοβ. Σε συνεχάριν ήδη. Θέλω να σε ευχαριστήσω όμως. Ευφυΐα και τεχνογνωσία έδωσες συνέβαλε με πολιτική αποφασιστικότητα στα πλαίσια ευρωπαϊκού πνεύματος εργασία μας. Το εκτιμούμε τα μάλα. Και εγώ και οι συνάδελφοι. Χαίρομαι ότι κάποια τα στοιχεία και τη δημόσια οπτική, την ευρωπαϊκή οπτική γωνία θα την φέρεις και στο Εθνικό Υπουργείο Οικονομικών. Όλοι μας ε, πρέπει να σου πούμε θα μας λείψεις. Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια εκ νέου για τη νέα σου θέση, τα νέα σου καθήκοντα. Συγχαρητήρια και τη δουλειά που έκανες εδώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Να διαβάσω το χρονοδιάγραμμα τώρα, το πρόγραμμά μας. Α, να το. Με επιφύλαξη, επίτευξη συμφωνίας. Καταρχήν η ψηφοφορία προβλέπεται για 21 Ιανουαρίου. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Επιτρέψτε μου να πάω στα σημεία 5 και 6. Καλωσορίζω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κ. Ντομπρόφσκης και τον Επίτροπο, τον κύριο Μοσκοβισή. Είναι έκτακτος οικονομικός διάλογος. Συγχωνεύουμε τρία θέματα. Τον τακτικό οικονομικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περί του φθινοπορεινού αυτού πακέτου. Έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και το σχέδιο εκθέσεως για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αποφασίσαμε επίσης να προσθέσουμε και νομική βάση. Άρθρο 7.3 του κανονισμού 473 του 2013 για να συζητήσουμε και την κατάσταση της Ιταλίας. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αρνητική γνωμοδότηση όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού, το προσχέδιο προϋπολογισμού και ζητήθηκε και αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού, δεν αναθεωρηθήκε, οπότε χρειάστηκε να ζητηθεί νομική άποψη για τον προϋπολογισμό, του σχέδιο προϋπολογισμού. Έχουμε λοιπόν καθήκον και προνόμιο, σύμφωνα με το ΤΟΥΠΑΚ, να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει ε, για την ιδιαίτερα αυτή δύσκολη οικονομική κατάσταση. Εστιαζόμενοι από αυτού. Δεν είναι μόνο συζήτηση περί Ιταλίας, γενική συζήτηση για το εξάμεινο είναι, αλλά θέλαμε να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Σύντομο σχόλιο από αυτό. Νομίζω ότι είναι θετικό το ότι λαμβάνει η χώρα διάλογος. Είναι προφανές ότι διατάξει περί ευελίξεως του Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αφορούν τα κράτη-μέλη όλης της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Αν η παρούσα κυβέρνηση θέλει να κινηθεί εντός αυτού του πλαισίου, αυτό θεωρείται θετικό και ευπρόσδεκτο. Θα εξετάσουμε προσεκτικότατα. Όμως το θέμα θέλουμε όλα να γίνουν στα πλαίσια του πνεύματος της νομοθεσίας. Δεν είναι μόνο θέμα αν είναι δυνατόν να υπάρχει ευελιξία, αλλά πρέπει η ευελιξία να παρέχεται εντός των κανόνων. Αυτό θα εξετάσουμε προσεκτικά στο επόμενο στάδιο του διαλόγου. Τώρα ήρθε η στιγμή να δώσουμε το λόγο στους επιτρόπους. Πρώτος αντιπρόεδρος ο κ. Ντομπρόφσκης έχει το λόγο. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Ρομπέρτο. Ε, αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την φθινοπορεινή δέσμη μέτρων στις 21 Νοεμβρίου. Θα ξεκινήσει το 2019 στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η οικονομία της Ευρώπης μπαίνει σε έκτο συνεχόμενο χρόνο ανάπτυξης. Η απασχόληση είναι σε, ε, σε άνοδο και υπάρχει γενικότερη ανάπτυξη. Αυτό δείχνει ότι η στρατηγική μας που βασίζεται σε τρεις προτεραιότητες, τις επενδύσεις, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική έχει αποτέλεσμα. Όμως υπάρχουν ορισμένες χώρες ε, όπου φαίνονται ακόμα οι επιπτώσεις ε, της ε, κρίσης. Η διόρθωση των μακροοικονομικών ανισοτήτων ε, συνεχίζεται, όμως ε, παραμένουν κάποια προβλήματα. Σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν ακόμα υψηλά επίπεδα χρέους, υπάρχουν ακόμα χαμηλά ποσοστά απορρόφησης και κάποια κράτη-μέλη ακόμα έχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας ή ε, από την άλλη έχουν έλλειψη εργοτικού δυναμικού θα σας ενημερώσω περισσότερο κατά την παρουσίαση του μηχανισμού ετοιμότητας. Έπειτα παραμένουν κάποια άλλα ζητήματα όπως ε, περιβαλλοντικά κτλ. Η μόνη λύση είναι να δημιουργηθεί περισσότερη ευημερία, να δοθεί όθηση στην στασιμότητα της αγοράς εργασίας σε ορισμένους ε, κλάδους και σε ορισμένες περιφέρειες υπάρχει ανισότητα εισοδηματική η οποία εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής ε, ακμής, όμως δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα προβλήματα και δεν μπορούμε επίσης να γνωρίσουμε το ότι η ευκαιρία που έχουμε δεν, για περισσότερη ανάπτυξη δεν θα κρατήσει για πάντα. Χρειάζεται να αυξηθεί η παραγωγικότητα σε εθνικό επίπεδο και, σε, ε, και να γίνουν περισσότερες καλές επενδύσεις, καθώς επίσης ε, και να δημιουργηθούν δημοσιονομικές αποθέματα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται ενίσχυση της ε, νομισματικής ε, οικονομικής ένωσης. Ε, συζητήθηκε ήδη η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, όμως ακόμα περιμένουμε να έρθουμε σε συμφωνία για άλλα θέματα όπως τη δημοσιονομική σταθεροποίηση και άλλα. Και αύριο στην συζήτηση στην Ολομέλεια θα έχουμε ελπίζω περισσότερα ε, καλά νέα. Τώρα γνωρίζω ότι η Επιτροπή σας καταρτίζει μια έκθεση για την ετήσια έκθεση ανάπτυξης, ε, γι' αυτό λοιπόν θα περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον ε, να τη διαβάσω ενίσχυση των ε, κεφαλαιογορών πολλές φορές συνοδεύεται από πρόσθετο κόστος. Χρειάζεται λοιπόν ε, να ενισχύσουμε τα προγράμματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει εξατομικευμένη στήριξη στα κράτη-μέλη που τη χρειάζονται. Για το 2019 έχουμε λάβει πάνω από 600 αιτήσει στήριξης και δεδομένης της ε, αύξησης του προπολογισμού ε, η ζήτηση έχει αυξηθεί κατά 100%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στήριξη μέσω εμπειρογνωμοσύνης, ε, όμως τα κράτη που θα ζητήσουν στήριξη θα λάβουν επίσης και οικονομική στήριξη. Ο δικός σας ρόλος είναι να προχωρήσετε και να ολοκληρώσετε το την έγκριση του προγράμματος για την ε, δημοσιονομική σταθεροποίηση. Περνάμε τώρα στις συστάσεις για την Ευρωζώνη. Η πρότασή μας εστιάζει σε ορισμένους βασικούς τομείς για την σωστή λειτουργία της Ευρωζώνης. Ζητά πολιτικές που θα ενισχύουν την ε, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα που θα ενισχύουν την συμμετοχή στην αγορά εργασίας και θα μειώσουν το ιδιωτικό χρέος και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, ε, ζητά μείωση του χρέους και δημιουργία αποθεμάτων για την αντιμετώπιση κινδύνου. Είναι καιρός ε, λοιπόν ε, για δράση. Αυτό είναι το μήνυμα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ε, Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ε, προπολογισμό. Έχουμε δημοσιεύσει τις εκθέσεις μας. Για πρώτη φορά όμως η έκθεση είναι για ε, τη συνολική Ευρωζώνη. Η Ελλάδα έχει καταθέσει το δικό της σχέδιο που συνάδει με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Χρειάζεται όμως να ε, πιάσει τους στόχους για να συνεχίσει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Αλλά ο συνάδελφός μου θα σα ενημερώσει επ' αυτού. Καμία χώρα τώρα δεν προβλέπεται να έχει έλλειμμα πάνω από το 3% του ΑΕΠ από την ε, εισαγωγή του ευρώ. Τα πράγματα φαίνονται λοιπόν καλά ε, ονομαστικά. Στην πράξη όμως είναι κάπως διαφορετικά. Η εφαρμογή ε, του προϋπολογισμού θα μας οδηγήσει σε αρκετές δυσκολίες, ιδιαίτερα για τα κράτη που έχουν ε, μεγάλο χρέος. Στην Ιταλία προβλέπεται επιδίνωση της ε, διαρθρωτικής ισορροπίας της. Η Αυστρία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Κύπρος μεταξύ άλλων είναι δέκα χώρες οι οποίες ε, έχουν συμμορφωθεί πλήρως. Η Εστονία, η Λατονία και η Σλοβακία έχουν συμμορφωθεί μερικώς ε, και οι υπόλοιπε, το Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Σλοβενία έχουν ελλειπή συμμόρφωση. Τέλος, δύο λόγια για την Ιταλία. Ήταν πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να ζητήσει από κράτος μέλους να ε, θεωρήσει το σχέδιο προϋπολογισμού. Το δημοσιονομικό σχέδιο της Ιταλίας έχει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τις συστάσεις του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο έκανε σύσταση στην Ιταλία να μειώσει το διορθωτικό λίμα στο 0,06% του ΑΕΠ, όμως εμείς βλέπουμε μια αύξηση του ελλείμματος κατά 1% του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια έπρεπε να επανεξετάσουμε την συμμόρφωση της Ιταλίας ε, με την αναδιάρθρωση χρέους τα περασμένα έτη δεν είχαμε προτείνει κάποιες αλλαγές στην ε, διαδικασία, μια που η Ιταλία ε, διασφάλιζε πως υπήρχε ευρύτατη συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τώρα όμως που δεν υπάρχουν αυτές οι διασφαλίσεις και μάλιστα δεν υπάρχει καν ε, ως στόχος για το επόμενο έτος, το άρθρο 126.3 αναφέρει ότι θα πρέπει να, με τις δεδομένων τούτων να θεωρείται ένα κράτος ως εμείς συμμορφούμενο και να ε, ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Η αξιολόγησή μας έχει ε, τύχει στήριξη και από το Eurogroup και από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν αφήσει τις ε, ελπίδας μας στην κυβέρνηση της Ιταλίας έτσι ώστε να αλλάξει αυτό και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις. Χρειάζεται όμως να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές σε ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η εμπειρία μας ε, δείχνει ότι το, το υψηλό χρέος δεν επιφέρει ανάπτυξη, αντίθετα κάνει την οικονομία πιο ευάλωτη. Επίσης η δημοσιονομική πολιτική έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Ήδη έχουμε αποδείξεις για αυτό για το επόμενο έτος, ότι το δημοσιονομικός σχεδιασμός ε, έχει άμεση σχέση ε, με την εμπιστοσύνη πολιτών και επενδύσεων. Πιστεύουμε πως η συμμόρφωση είναι όχι μόνο προς το συμφέρον της Ιταλίας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν μετά από τις συζητήσει που θα γίνουν και το αποτέλεσμα αυτών. Τώρα θα ζητήσω από τον αγαπητό Πιέρ να ε, συνεχίσει την παρουσίαση για τα επιμέρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Μπάλτη. Όπως είπε και ο μπάλτη, αυτός ο οικονομικός διάλογος μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου είναι ύψιστης της σημασίας για την διαφάνεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ξέρετε ότι προσδίδω μεγάλη σημασία σε αυτό. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό εξάμεινο, το τελευταίο ευρωπαϊκό εξάμεινο πριν από τις εκλογές του Μαΐου του 2019 και θα πρέπει να δούμε πώς ορίζεται η κατάσταση και με βάση την Ένωση, με παράδοξο Η Ευρωζώνη έχει θετικό πρόσημο. Η ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη υφίσταται, αν και κάπως επιβραδυμένη, αλλά στην Ευρώπη υπάρχουν ανισότητες οικονομικές, αλλά και πολιτικές, καθώς και πολιτικοί κίνδυνοι που γνωρίζουμε. Στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα ήθελα να μιλήσω για το μηχανισμό ειδοποίησης. Πρόκειται για μια διαδικασία, μακροοικονομική διαδικασία και η Επιτροπή αποτιμά τους κινδύνους. Τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους εκινήθηκε αυτή η διαδικασία για να διορθωθούν οι μακροοικονομικές ανισότητες και για να ορίσει τις ευάλωτες ζώνες σε ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα όπου ο ιδιωτικός τομέας φαίνεται ιδιαίτερα ε, άνισος. Επίσης, η τιμή της στέγης καθώς και οι μισθοί γνωρίζουν μεγάλες ανισότητες. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να εξετάσει εις βάθος την κατάσταση 11 κρατών όπου υπάρχουν μεγάλες ανισότητες. Ε, Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία ε, και άλλες τρεις χώρες. Δύο χώρες εξετάζονται ιδιαίτερα, η Ρουμανία δηλαδή, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι ως προς την ανταγωνιστικότητα και η Ελλάδα την ε, κατάσταση της οποίας θα αποτιμήσουμε μετά την λήξη του τρίτου μνημονίου και θα δούμε πώς ορίζεται η κατάσταση αναχώρα. Αυτό θα γίνει στις αρχές του 2019. Θα ήθελα να σας πω τα συμπεράσματα του δημοσιονομικού ελέγχου συμπληρώνοντας αυτά που είπε ο Βάλτης. Η πλειοψηφία των κρατών μελών ακολούθησαν την ε, ανάκαμψη του δημοσίου τομέα και το έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι κάτω από το 1%, δηλαδή 0,6 και 0,8%. Είχαμε ένα 30% επίσης Όσον αφορά το χρέος, θέλαμε να περάσουμε σε ένα χρέος κάτω από το 60% του ΑΕΠ. Η Γερμανία και η Ολλανδία θα χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο για τις κατάλληλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ζητούσε αυτές τις διορθώσεις και χαιρόμαστε γιατί έγιναν. Βεβαίως, το 19 δείχνει ότι πολλές χώρες δεν δείχνουν επάρκεια. Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία δείχνουν ότι δεν ανταποκρίνονται στις δημοσιονομικές ανάγκες. Μιλάμε λοιπόν για μία περίοδο ανάπτυξης, αλλά αυτές οι χώρες θα πρέπει να μειώσουν το δημόσιο χρέος. Θα ήθελα να επιμείνω σε δύο περιπτώσεις της Ιταλίας και της Ελλάδας. Καταρχήν, όσον αφορά την Ιταλία, η ανάλυση μας δείχνει ότι υπάρχει κίνδυνος μη συμμόρφωσης, πολύ σοβαρός κίνδυνος σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μετά τις 20 Νοεμβρίου, ο διάλογος με τις Ιταλικές Αρχές συνεχίζεται επικοδομητικά και εντατικά. Ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, συναντήθηκε με, τον, ε, με τους Κόντε και Τρία και στον Buenos Aires επίσης είχαμε θετικές συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό Κόντε και τον Υπουργό Οικονομικών Τρία και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα. Εδώ και δύο εβδομάδες υπάρχει ένας διαφορετικός τόνος και διάθεση συνεργασίας από τις Ιταλικές αρχές, κάτι το οποίο χαιρετίζω. Οι Ιταλικές αρχές θέλουν να μειώσουν το έλλειμμα το 2019 και έχουν γίνει και πολλές ε, πολιτικές ανακοινώσεις επί του θέματος. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν απτές δεσμεύσεις με αριθμητικά στοιχεία για να κινηθούμε όπως πρέπει, για να αλλάξουμε την ανάλυση μας. Η Επιτροπή έδειξε πάντα ευελιξία έναντι της Ιταλίας για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, για την κυκλική οικονομία, για την ασφάλεια και τις φυσικές καταστροφές. Μιλάμε για 30 δις συνολικά. Και επίσης ε, χρησιμοποιήσαμε κάθε περιθώριο που διαθέταμε. Όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους κανόνες του συμφώνου που πρέπει να σέβονται όλα τα κράτη-μέλη και δεν μπορούμε να προβαίνουμε σε παρεκκλήσεις, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται ε, στους κανόνες «Pacta sunt servanda». Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει τα επόμενα ε, νομικά βήματα στα πλαίσια του, ε, της δραστηριότητας του Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια του υπερβολικού ελλείμματος για να εκινήσουμε την δέουσα διαδικασία. Θα πρέπει να προωθήσουμε τον διάλογο και να προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα. Αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο και στο μεταξύ υπερασπιζόμαστε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, δημοσιονομικούς κανόνες, και φυσικά υπάρχει και το χρονόμετρο, το οποίο δεν πρέπει να αγνοούμε Ως προς την Ελλάδα, η Επιτροπή παρακολούθησε την κατάσταση της Ελλάδας. Υπάρχουν ορισμένες ε, καθυστερήσεις, αλλά κανένα τρένο δεν φτάνει στην ώρα του. Η Ελλάδα έχει επιτύχει μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εξαμήνου και βλέπουμε ότι θα υπάρχει πρωτογενές ε, πλεόνασμα γύρω στο 3,6% του ΑΕΠ, έτσι ώστε να μην γίνουν περικοπές στις συντάξεις το 2019 και 2020. Αυτό το επικύρωσε και το Eurogroup και ο επόμενος προϋπολογισμός θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Θα υπάρχει και μία ενισχυμένη αξιολόγηση και εποπτεία. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο γιατί υπάρχουν άνισα αποτελέσματα από τον ένα τομέα στον άλλο. Οι ελληνικές αρχές γνωρίζουν πολύ καλά τι ακριβώς πρέπει να κάνουν για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Γιατί αυτό θα ορίσει και την επόμενη δόση της τάξης του, των 750 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά θα πρέπει να καταβληθούν και προσπάθειες για να έχουμε ένα success story. Έτσι ώστε η Ελλάδα μέσα στα πλαίσια της ε, εθνικής κυριαρχίας να προωθήσει τις οικονομικές και κοινωνικές ε, συνιστώσεις για να μπορέσει να φτάσει σε μια απτή ανάπτυξη. Ευχαριστώ τον Βάλτης Ντομπρόφσκης και τον Πιέρ Μοσκοβισή. Να υπενθυμίσω στους φιλοξενούμενους μας και τους συναδέλφους ότι στις 9 ακριβώς θα πρέπει να ψηφίσουμε οπότε θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός όσον αφορά το χρόνο και θα πρέπει ο καθένας να μιλάει για 4 λεπτά. Διαφορετικά θα προλάβουμε τις ψηφοφορίες μας στις 9. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο σας. Υπήρξατε σαφέστατοι. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Δίκαιη προσπάθεια για διάλογο, για επικοδομητικές λύσεις. Η διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος θα ήταν αρνητική εξέλιξη για την Ιταλία. Είναι δίκαιο που ισότιμα παρέχεται η ε, ευελιξία, ανεξάρτητα από το αυτή είναι η χώρα μου αμερόληπτα. Αλλά και η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι κάθε παιχνίδι έχει και το όριό του και θα πρέπει να δώσει αξιόπιστα στοιχεία και να αναλάβει υποχρεώσει. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτή η επικοδομητική προσέγγιση θα βοηθήσει και τις δύο πλευρές και θα σημειωθεί πρόοδο σε επόμενε ημέρες. Διότι μας τελειώνει και ο χρόνο. Ευχαριστώ εκ νέου για την επικοδομητική προσέγγιση που ακολούθησαν οι κύριοι Μοσκοβισί και Ντομπρόσκη. Πάμε στου ομιλητέ μα. Ο εισηγητή για το εξάμεινο. Ο κ. Βραντέκαλαρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω λίγο χρόνο να φορέσετε τα ακουστικά σας για να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Έχω δύο σχόλια. Θα αναφέρω τα σχόλιά μου στο τετράλεπτο για τη γύρανση του πληθυσμού. Θέλω να μιλήσω και για την Ιταλία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυξανόμενη γύρανση του πληθυσμού. Και νομίζω ότι χρειάζεται μακροπρόθεσμο όραμα. Καμιά φορά αυτό είναι δύσκολο να συμφιλειωθεί με νομοθετικές περιόδους συγκεκριμένες. Ο κ. Μοσκοβισή σωστά είπε ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα συζητήσουμε το θέμα πριν τις ευρωεκλογές πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για μια μακροπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων. Χρειάζεται δράση. Το κόστος της γύρανσης αυξάνεται συνεχώς και θα αυξηθεί ε, το πρόβλημα της επόμενης δεκαετίας από πλευράς περίθαλψης και συντάξεων. Αν θέλουμε να δούμε την αύξηση του πληθυσμού που πρέπει να καλύπτεται, έχουμε αλλαγή των πραγμάτων. Λιγότεροι θα πληρώνουν εισφορές και περισσότερες συντάξεις πρέπει να καταβάλλονται. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε απάντηση στο πρόβλημα. Διαφορετικά θα υπάρξει τεράστιος αντίκτυπος για τη βιωσιμότητα της οικονομίας των χωρών μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει γι' αυτό. Από καιρούς καιρών αναφέρεται το θέμα και έχει αναφερθεί ότι χρειάζεται ένα μελλοντικό σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια βήματα πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθηθούν για να αντιδράσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό ήταν το πρώτο, για την Ιταλία τώρα. Είδαμε διαμαρτυρίες την προηγούμενη εβδομάδα. Και δεν τονίζονται παρκώς, πιστεύουμε, οι επενδύσεις. Και υπάρχουν ανησυχίες για την Ιταλική οικονομία για το μέλλον. τα προβλήματα βαίνουν αυξανόμενα. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων επενδύσεων, αυτών που είναι περισσότερο ε, παραγωγικές επενδύσεις από ό,τι άλλες. Απάντηση. Κ. Ευχαριστώ για αυτές τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω από την πρώτη ερώτηση για τα μακροπρόθεσμα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και η γύρωση του πληθυσμού. Στη διαθροτική μεταρρύθμιση τονίσαμε ιδιαίτερα μεταρρυθμίσεις μακροπρόθεσμες του συνταξιδοτικού συστήματος, συστήματος προνοίας, ούτω ώστε τα συστήματά μας να είναι βιώσιμα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε και πάρκια των συντάξεων Ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στις συστάσεις αναχώρα, αυτό από τη μια πλευρά, και από την άλλη δεν θέλουμε να σταματήσουν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί, όπως βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες όσο πιο έγκαιρες γίνονται οι προσαρμογές, τόσο λιγότερο δραματική η φύση τους. Άμα έχουμε ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο σωστό για την Ιταλία και τις επενδύσεις. Όπως ξέρετε η Ιταλία είναι μια χώρα που έχει ωφεληθεί περισσότερο από τη συμπροματική ευελιξία που εφαρμόζεται βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Είναι από τις μεγαλύτερες χώρες δικαιούχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του σχεδίου Juncker, όπως λέγεται αλλιώ για επενδύσεις. των διαθωτικών ταμείων, των ταμείων συνοχής, έχει ευνοηθεί από όλα αυτά. Άρα υπάρχει περιθώριο επαρκών επενδύσεων. Πρέπει να δούμε ότι ό,τι γίνεται θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο δημοσιονομικά βιώσιμο. Πρέπει να αποφευχθεί αύξηση ε, των, του κρατικού χρέους και του, γενικά του χρέους. Δεν θα είναι τελευταία ερώτηση επί της Ιταλίας, οπότε πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πρέπει να είμαστε αυστηροί όσον αφορά τις χρονοθυρίδες. Περές. Το θέμα της Ιταλίας θέλω να θίξω. Όλοι και ο Επίτροπος Μοσκοβισή γνωρίζουν ότι αν πετυχαίνει κάτι κάποιο από τις Βρυξέλλε, χρησιμότερο είναι ο διάλογο και όχι οι κλειστές πόρτες. Το ότι μπήκαμε σε αυτή τη φάση σίγουρα είναι θετικό. Η πορεία που ακολούθησε η Ιταλία δημιουργεί ερωτηματικά. Κατά την άποψή σας, η σωστή πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η Ιταλία όχι απαραίτητα για να συμμορφωθεί με το Σύμφωνο σταθερότητα και Ανάπτυξης. Ούτε στα πλαίσια της Ευρωζώνης, αλλά για να βρει μια πορεία ανάπτυξης η Ιταλία που θα επιτρέψει στους Ιταλούς πολίτες να αναγνωρίσουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα και το ευρώ. Χωρίς να θεωρήσουν ότι είναι δώρα που θα φέρει μόνο ο Άι Βασίλης. Ποια είναι η άποψή για την πορεία τη Ιταλία, για την Ελλάδα. Μπορείτε να διευκρινίσετε κάποια πράγματα. Πώς ορίζονται νέε διευθετήσεις. Άλλαξε κάπως η κλίμακα. Περάσαμε από ένα πρόγραμμα. Δεν είναι πλέον υποπρόγραμμα. Έχουμε μια νέα διαδικασία που ξεκίνησε για πρώτη φορά. Εκεί εντάσσεται η Ελλάδα. Ποιες ρυθμίσεις οργανώσατε αυτό το μηχανισμό, αυτό το σύστημα που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Ο κ. Μοσκοβισή, δεν θα σχολιάσω αν είναι δικαιολογημένο ο χαρακτήρα ή όχι του συμφώνου. Έχει ένα, μια λογική το συμφωνώ. Το δημόσιο χρέο που είναι απόλυτο εκτός της οικονομίας, διότι στερεί κάθε, κάθε χώρα από την δυνατότητα ελιγμών για σωστές επενδύσεις, εμποδίστε το δημόσιο Έχει επίπεδο χρέος η Ιταλία 131% και η πορεία που παρουσίασε αρχικά δεν επιτρέπει τη μείωση του χρέους. Και την πορεία που ακολουθούν, ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν αργό ρυθμό, αλλά δεν τον ακολουθεί η Ιταλία το σχέδιο προπολογισμού θα οδηγούσε σε συνέχιση του αυξήσεως του δημοσίου χρέους. Με έναν προπολογισμό που οδηγεί σε μείωση του ρυθμού αναπτύξεως και στη φτωχοποίηση. Περιμένουμε τις δέουσες απαντήσεις από την Ιταλία για να αλλάξει πορεία. Δεν υπάρχει μαγικός αριθμός. Ε, αλλά θέλουμε να ακολουθεί η λογική του συμφώνου. Μία πορεία δηλαδή να θεσπιστεί που επιτρέπει τη μείωση του δημοσίου χρέους. Και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε το σωστό μονοπάτι που δεν θα στερεί την Ιταλική κυβέρνηση που έχει εκλεγεί νόμιμα από το δυνατότητα ελιγμών αλλά θα πρέπει οι επιλογές που κάνει η κυβέρνηση να συνάδουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Υπάρχει το μονοπάτι. Και έτσι θα μειωθεί το δημόσιο για την Ελλάδα. Αποτελεί αντικείμενο ενισχυμένης εποπτείας, αυξημένη εποπτείας. Φροντίσαμε αυτή η εποπτεία ενισχυμένη να μην είναι τέταρτο πρόγραμμα και καλυμμένο και οι λεπτομέρειες εποπτείας να μην αντιστοιχούν σε ένα, κρυμμένο, ένα κρυμμένο πρόγραμμα εποπτείας. Είναι, είναι εποπτεία όπως κάνουμε άλλα κάτι μέλη. Ενισχυμένο καθεστώς για να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις. Έχουμε τέσσερις εκθέσεις το χρόνο. Δύο έγιναν για να συμπέσουν με το στάδιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και πρέπει να σας πω ότι η πρώτη αυτή αποστολή ολοκληρώθηκε υπό τι καλύτερε δυνατέ συνθήκε. Η συνεργασία με τι ελληνικέ αρχέ ήταν άριστη. Και βλέπει να δούμε τι λειτουργήσε, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά και να αποτιμήσουμε τι απομένει να γίνει, τι πρέπει να κάνει ακόμα η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Καρολίνα Τάρη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης, κύριε Επιτροπέ, κύριε Μοσκοβισή, που ήρθατε εδώ για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων για ε, τον προϋπολογισμό των ε, κρατών μελών, ιδιαίτερα για την περίπτωση της Ιταλίας. Θα ήθελα να μιλήσω για την ε, δύσκολη στάση που και την αυστηρή μάλλον στάση που τήρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν δύσκολα τα πράγματα στο παρελθόν, όμως έχω κάποιες ανησυχίες για το πλαίσιο στο οποίο παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός της Ιταλίας. Ήταν διαφορετικά από ό,τι περίμεναν οι ίδιοι Ιταλοί πολίτες και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον ε, το ποσοστό του λίμματος, το 2,9%, λίγο κάτω από το 3%. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν έχει συζητηθεί αυτό το ποσοστό, αν έχουν συζητηθεί τα όρια αυτά, διότι ίσως θα έπρεπε να γίνει μια ουδέτερη αξιολόγηση. Επίσης, ο προϋπολογισμός της Γαλλίας, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος προϋπολογισμός, έχει ε, ποσοστό ελλείμματος 2,8% και θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως αυτό είναι εφικτό. Θεωρείται πως ο πρόεδρος Μακρόν θα υιοθετήσει μια προσέγγιση όπως αυτή της Ιταλίας, όπως αυτή άλλων χωρών, θα υπάρξει μείωση του ελλείμματος, Νομίζω πως ε, δεν θα έπρεπε να είμαστε ρηψοκίνδυνοι και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ερωτήσεις. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την Ιταλία. Αναφέρατε στο ονομαστικό έλλειμμα και όπως γνωρίζετε εδώ τα νούμερα διαφέρουν. Οι προβλέψεις ε, τη Ιταλία είναι 2,4%, οι οικονομικές προβλέψεις της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 2,9%, το ποσοστό δηλαδή που αναφέρατε κι εσείς. Όμως, ε, στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν μετράμε μόνο το ονομαστικό έλλειμμα. Το 3% όπω είπατε κι εσεί συνάδελφε δεν είναι ο στόχος. Αυτό που μετράτε είναι εάν ο προϋπολογισμός των κρατών μελών βρίσκεται σε ε, έναν κύκλο, σε μια κυκλική τάση και είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να συγκλίνουν προς έναν εξορθολογισμένο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του οικονομικού του κύκλου. Αυτή είναι μία απλουστευμένη βέβαια προσέγγιση. Μετά, αναφερθήκατε στην περίπτωση της Γαλλίας. Ας κάνουμε λοιπόν μια σύγκριση. Η Ιταλία και η Γαλλία έλαβαν συστάσεις έτσι ώστε, το 0, έτσι ώστε να σημειωθεί 0,6% διαρθρωτική βελτίωση. Η Γαλλία έχει σημειώσει διαρθρωτική βελτίωση 0,2% σύμφωνα με τις ε, δικές τους προβλέψεις. Η Ιταλία σύμφωνα με τις προβλέψεις κυβέρνησης έχει επιδείνωση 0,4%. Βλέπουμε λοιπόν πως πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις και ως τελείως διαφορετικές πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επίσης, το ονομαστικό έλλειμμα της Γαλλίας φέτος είναι όντως υψηλότερο και είναι ένα από τα μεγαλύτερα δεδομένων των ε, αλλαγών στην ε, πολιτική φορολόγησης. 1,9%. Επίσης, παρακολουθούμε στενά την εξελίξεις και εξετάζουμε το ενδεχόμενο επιβολής νέων μέτρων. Αυτό βέβαια θα ε, ανακοινωθεί στο μέλλον όταν έχουν εξεταστεί όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες. Πρώτα όμω πρέπει να σημειωθεί πρόοδο και μετά να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Θα ήθελα κι εγώ να προσθέσω κάτι σε σχέση με τη σύγκριση Γαλλίας-Ιταλίας. Οι κανόνες είναι ίδιοι για όλους. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση ούτε περιθώρια ερμηνείας. Σβέν Γκίγκολτ. Ευχαριστώ. Η κατάσταση ως προς την Ιταλία δεν είναι καθόλου απλή. Από τη μία πλευρά οι κανόνες του Six Pack καθώς και άλλοι είναι πολύ προκυκλικοί και κάναμε ουσιαστικά λάθη όταν φτάσαμε στο συμβιβασμό των έξι νομοθετημάτων. Επίσης, δεν μπορεί να υπάρχει νόμισμα και προϋπολογισμός χωρίς κανόνες. Το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ιταλίας ε, είναι ε, ένας ε, προϋπολογισμός ψευδοοικονομικών κινήτρων γιατί για τα επιπρόσθετα ευρώ που δαπανώνται θα πρέπει να καταβληθεί δύο φορές ο τόκος καθώς και τα ασφάλιστρα επενδύσεων. Άρα δεν υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Για να είμαστε σαφείς και η Επιτροπή δεν απάντησε σαφώς, με σαφήνεια. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα νομικής ανασφάλειας, διότι εσείς βασίσατε την παρέμβασή σας όχι στο έλλειμμα, αλλά στα κριτήρια του χρέους. Όμως θεωρήσατε ότι τα καλύπτεται επαρκώς εάν ευθυγραμμίζεται και το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Όμως, αυτό δεν ήταν καθόλου συνειδητό και να, για να το πω πολιτικά. Δεν πιστεύετε στο κριτήριο του χρέους για τις χώρες με υψηλό χρέος, γιατί αν υποχρεώσετε την Ιταλία να μειώσει το χρέος κατά 3,5% του ΑΕΠ ετησίως, τότε θα σκοτώσετε την Ιταλική οικονομία άρα δεν εφαρμόσατε το κριτήριο του χρέους και τώρα βασίζετε τη νομική σας προσφυγή σε αυτό το κριτήριο. Άρα τα έξι νομοθετήματα έχουν σοβαρές ελλείψεις. Μπορείτε να ανταποκριθείτε στις επικρίσεις ως προς τα έξι νομοθετήματα που έχουν πολλά νομικά χάσματα και είναι πάρα πολύ δυσνόητο αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει να βρεθούν άλλοι πιο ευνόητοι κανόνες. Σε σχέση με τη Γερμανία, το πλεόνασμα της Γερμανίας στις μακροοικονομικές ανισότητες είναι, ευραίος, είναι κάτι το ευρέως γνωστό πότε θα λάβετε σαφή δράση κατά, τον, ε, κατά του πλεονάσματος της Γερμανίας. Διαφορετικά, εσείς δημιουργείτε ανισότητες στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θα πρέπει λοιπόν να, λάβετε, να αναλάβετε δράση έναντι όλων των ανισοτήτων. Μοσκοβισή. Η συζήτηση ε, επί των κανόνων δεν αποτελεί ταμπού για την Επίτροπη αυτή. Κάνουμε επανεκτιμήσεις συνέχεια. Μπορεί οι κανόνες να είναι πιο απλοί και ίσως θα μπορούσαν να διασαφινιστούν. Γιατί υπάρχει μία ενιολογική βάση που είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Όμως, τι ζητήσαμε από την Ιταλική κυβέρνηση στην επιστολή μας ως προς τη γνωμοδότηση και το follow-up. Μιλήσαμε για το διαρθρωτικό έλλειμμα, για το δημόσιο χρέος και για την ανάπτυξη. Και η διασύνδεση των τριών είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός αυτός δεν είναι ε, αρκετά ακρίβης ως προς το χρέος και δεν μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη ανάπτυξη λόγω του σκέλους των επενδύσεων και της απόκλησης αυτής που προϋπάρχει, αν λάβετε υπόψη το σύνολο των κανόνων. Καθίσταται σαφές ότι έχει μεγάλη σημασία το κριτήριο του χρέους. Γι' αυτό προωθούμε και τον εν διάλογο και δεν προτρέχω. Δεν φτάνω σε συμπεράσματα. Θέλουμε να προωθήσουμε έναν διάλογο που να οδηγήσει σε λύσεις ημεριζόμενες και από τις δύο πλευρές για να φτάσουμε σε συμπεράσματα ή δυνατόν αλλά συνεργαζόμαστε και ως προς το διάλογο και την προετοιμασία για να δούμε ποια θα είναι η έκβαση καταρχήν του διαλόγου. Στην περίπτωση της Γερμανίας έχουμε δύο διαδικασίες αναχείρας, αλλά δεν είναι ταυτόσιμες. Η μία είναι απόλυτα ακριβής, με μηχανισμούς με πιθανές κυρώσεις και το άλλο σκέλος είναι εντελώς διαφορετικό. Σήμερα όμως για πρώτη φορά όλες οι χώρες τείνουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και η Γερμανία κάνει το ίδιο ως προς το χρέος και καταβάλλεται η προσπάθεια χρήσης των πλεονασμάτων για επενδύσεις για την μείωση των ε, διαρθρωτικών ανισοτήτων. Θα κάνουμε μία εις έρευνα σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και την Γερμανία, και μετά θα υποβάλουμε προτάσεις στα πλαίσια του εξαμήνου. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους ε, κύριους επιτρόπους που ήρθατε εδώ για τον διάλογο αυτό. Δεν θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για την Ιταλία, αλλά ε, θα ήθελα να πω το εξής. Ε, η Μηχανισμός σταθερότητας, ο ρόλος του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μία ανακοίνωση όπου αναφέρεται στην ενίσχυση του ευρώ. Με την ανακοίνωση αυτή δημιουργούνται κάποιες προϋποθέσεις για την ενίσχυση ε, του ευρώ, για αύξηση ε, του ισολογισμού έναντι των, ε, του υπόλοιπου κόσμου, αλλά αυτό σημαίνει και αύξηση του πλεονάσματος. Ε, εμείς όμως ε, δεν έχουμε ακόμα κάποια διαδικασία αντιμετώπισης της περίπτωσης χωρών με υπερβολικό πλεόνασμα. Όπως είπε και ο κύριος Γκίγκολτ, υπάρχουν χώρες με υπερβολικό μεγάλο πλεόνασμα, οι οποίες δημιουργούν αυτές τις ε, ανισορροπίες. Στην αρχή χρησιμοποιήσαμε τον ε, μηχανισμό σταθερότητας ε, και του δώσαμε το ρόλο του πιστωτή, του δανειστή. Τώρα βλέπουμε πως αυτή η τακτική επεκτείνεται, χρειάζεται όμως πράγματι κάτι τέτοιο και οι πιστώσεις δεν θα έπρεπε να είναι ε, εφικτό να αποπληρωθούν. Διότι στο τέλος ο φορολογούμενος είναι αυτός που ε, αναλαμβάνει και απομίζεται το κόστος αυτού του δανεισμού. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ερωτήσεις. Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ανακοίνωση. Αφορούσε την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ εξετάσαμε τους τομείς εκείνους τους οποίους μπορούσαμε να το πετύχουμε στην πράξη. Στον τομέα των πληρωμών, Φερρυπίν, του διεθνούς εμπορίου και εκεί κάναμε συστάσεις απευθυνόμενοι προς τα κράτη-μέλη όσον αφορά το εμπόριο στον τομέα της ενεργείας, χρήση του ευρώ σαν νόμισμα αποθεματικού και για το ισοζύγιο τρεγουσών πληρωμών η χρήση του ευρώ ως νόμισμα για διεθνές αποθεματικό. Διότι η διθεσιμότητα πόρων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν διεθνή αποθεματικά νομίσματα εκτός της ε, Ευρωζώνης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να χρησιμοποιείται το ευρώ για αποθεματικό. Στην ανακοίνωση δεν έχουμε συγκεκριμένα βήματα που προτείνουμε. Αυτό θα γίνει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως είπε ο Επίτροπος Μοσκοβισή. Στα πλαίσια της διαδικασίας μακροοικονομικών διαφορών, όπου χώρες με μεγάλα πλεονάσματα, τον όπως είναι η Ολλανδία και η Γερμανία, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των μακροοικονομικών ανισορροπιών και είναι κάτι που καλύπτεται σε αυτό το εξάμεινο και θα γίνει δελεχής ανάλυση των οικονομικών τους. Όσον αφορά το θέμα αυτό του Ταμείου Εξυγένσης και Ρευστοποίησης, και πώς μπορούν οι τράπεζες να επιστρέψουν τους πόρους που χρησιμοποιούνται από το Ταμείο Εξεγίανσης, που παίρνουν από το Ταμείο Εξεγίανσης. Έχουμε γι' αυτό τον ενίο φορέα εξυγένσης. μια τράπεζα που θεωρείται ότι είναι συστημικά σημαντική και θα πρέπει να διασωθεί και να εξυγενθεί για το κοινό συμφέρον, υπάρχει ένα σχέδιο εξυγένσης. Αυτό συνεπάγεται μεσοπρόθεσμη ε, βιωσιμότητα της τράπεζας και αποφεύγουμε τη χρήση των χρημάτων του φορολογωμένου Γι' αυτό έχουμε τον μηχανισμό, ενίο μηχανισμό εξυγένσης και το Ταμείο Εξυγένσης, το οποίο καλύπτεται από εισφορές του τραπεζικού τομέα. Θα χρησιμοποιηθεί για αυτό σκοπό. Και συζητούμε και το δημοσιονομικό μέσο στήριξης αυτού του Ταμείου. Η ερώτηση είναι τι γίνεται αν ξεμείνει από χρήματα το Ταμείο Εξυγένσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να επιταχύνουμε τη δημιουργία ενός οικονομικού μέτρου ασφαλείας για τη στήριξη του Ταμείου και για τη μείωση του κινδύνου του αντιμετωπίζει τραπεζικού τομέα. Αυτοί οι φορείς χρησιμοποιούνται, θα χρησιμοποιηθούν σαν ένα δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση προβληματών. Ευχαριστώ πολύ. Η Λάουρα Τζέα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, ευχαριστώ για την προσοχή που επιφυλάσσετε στην Ιταλία. Αλλά μέσω θέλω να κάνω κάτι ξεκάθαρο. Δεν δέχομαι και δεν συμμερίζομαι αυτό που υπονοείται, λέγοντας ότι η χώρα μου είναι μια χώρα που σπαταλάει πολλά. Το δημόσιο χρέος της Ιταλίας δεν είναι αποτέλεσμα ε, σε αυτό οφείλεται στις εσφαλμένες πολιτικές που εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και την αυξανόμενη δαπάνη για τους στόκους. Υγείτο η Ιταλία για την οικονομική ανάπτυξη ψηρά ετών. Μια δύναμη Ιταλία που δεν μπορεί πλέον να αναπτυχθεί, αυτό θα έπρεπε να ανησυχεί την Ευρώπη, να είναι πηγή ανησυχιών για την Ευρώπη. Θα έπρεπε να είναι μια πηγή ανησυχιών για την Ευρώπη μια δύναμη Ιταλία. Το ΑΕΠ αποταλμώνεται και αυξάνεται το χρέος. Αυτά είναι στοιχεία που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Και χρειάζεται αλλαγή ρυθμού. Το ζητούν οι πολίτες και το εφαρμόζει η παρούσα κυβέρνηση και θα πρέπει να υποστηρίξετε κι εσείς. Και η πεποίθησή μας είναι ότι η ενδυμική μείωση του ΑΕΠ βασικά οφείλεται στις πολιτικές λιτότητας που απέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησαν ένα φαύλο κύκλο και ασταμάτητη αύξηση ε, του συσχετισμού χρέους ΑΕΠ. Όπως υπεθυμίστηκε και από, άλλο, από διάφορα βραβεία Νόμπελ, από το Στίγκλης ξεκινώντα, η αύξηση της ζήτησης είναι στους παραγόντες που μπορεί να αυξήσει τον πλούτο που παράγει μια χώρα. Ο ελιγμός που προτείνει η Ιταλία, που προτείνει η παρούσα κυβέρνηση, είναι ελιγμό ε, αυξητικός, επεκτατικό Και χάρη και σε στιγμή αύξηση του δημόσιου χρέους θα μπορέσουμε να, να ζωγονίσουμε την οικονομία. Να πούμε όχι στη λιτότητα δεν σημαίνει ότι είμαστε ανευθυνοί, σημαίνει ότι αλλάζουμε δρόμο. Αν αυτός ο δρόμος που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα φαίνεται ότι είναι αδιέξοδο. Οι ιδέες μας έχουν την υποστήριξη των πολιτών. Και επιτρέψτε μου να σας πω με κάποια υπερηφάνεια Διαφορετικά από τι κυβερνήσει των βασικών χωρών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, θα έλεγα ότι η κυβέρνηση Κόντε απολαμβάνει τη συνενέσεω του 60% των Ιταλών πολιτών. 60% την υποστηρίζει. Και αυτό κάνουμε. Η εφαρμογή του ε, εισοδήματο ηθαγένεια, που είναι και κίνητρο για απασχόληση, είναι πραγματική διαθωτική μεταρρύθμιση τη αγορά-εργασία. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του ελιγμού αφιερώνεται στην επαναπρόθεση των δημοσίων επενδύσεων και αυτές που έχουν στόχο τις υποδομές που στα πλαίσια για της τεχνολογικής επιστημονικής έρευνας. Είμαστε υπερήφανοι για, αυτή την, για αυτόν τον ελιγμό. Αγαπητοί Επίτροποι, ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ιταλικής Κυβερνήσεως είναι κομβικό σημείο. Σας καλούμε ε, να κάνετε να επικρατήσει κοινή λογική. Όπως ακούσαμε και απόψε, μην κολλάτε στα δεκαδικά στοιχεία όταν ένας ολόκληρος ε, λαός απαιτεί αλλαγή. Ευχαριστώ. Ο Μοσκοβίση. Ευχαριστώ κυρία Βουλευτή. Είναι κατανοητή η πολιτική που ακολουθείτε, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να υπονομεύσει, αμφισβητήσει τις πολιτικές που επιλέγονται ή τις την άποψη και την εκλογή του Ιταλικού λαού που εκλέγει την κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι θέμα. Ανεξάρτητα από την ερμηνεία που δίνουμε στην αύξηση του χρέους, το ύψος του είναι πρόβλημα και για την Ιταλία και την Ευρωζώνη. Και είναι αποφασιστική σημασία αυτό. Για την γνωμοδότηση τη Επιτροπή Οικονομική Ομοσπονδιακή που ανεκρίθηκε από το Eurogroup. Η Ευρωζώνη είναι χώρος αλληλέγγυο, μην το λησμονείτε. Ή όπως έλεγε ο Γκίγκολτ, χωρίς κανόνες δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Πρέπει να εφαρμόζονται από όλου οι κανόνες τη Ευρωζώνη. Τρία σχόλια. Όσον αφορά το βασικό θέμα. Το θέμα του διαλόγου και της ανάπτυξης από την άλλη. Δεν μπορούμε να λέμε ότι επιβάλαμε στα τυφλά μια λιτότητα στην Ιταλία. Όπως υπενθύμησα προηγουμένω, και όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος, αυτή η Επιτροπή χρησιμοποίησε κάθε διαθέσιμη ευελιξία στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ανάπτυξης κάθε ε, ευελιξία, επενδύσεις, ε, κυκλικός χαρακτήρας, φυσική καταστροφές, ε, υπέρ της Ιταλίας. Και η Ιταλία ήταν η μόνη χώρα που βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση. Και είμαστε σε βαθμό να αποδείξουμε ότι αυτή η ευελιξία αντιπροσώπευε 30 δις ευρώ. 45 ε, δις ευρώ από το Εθνικό Ταμείο και 10 δις από αλλού προβλέφτηκαν. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι εμποδίσαμε την Ιταλία από το να κάνει επενδύσεις. Δεν μπορεί να λέγεται αυτό. Όλοι οι οικονομολόγοι φρονούν ότι το βασικό αίτιο της αδυναμίας της ανάπτυξης οικονομίας στην Ιταλία οφείλεται στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Και μόνο ρυθμίσεις στον τομέα της ανταγωνιστικότητας θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Όσον αφορά την ανάπτυξη, βλέπουμε ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα. Υπάρχει αποτελμάτωση της ανάπτυξης. Έχουν ανησυχίε οι οικονομικοί φορείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι διεθνείς οργανισμοί δεν έχει την ίδια πρόβλεψη ανάπτυξης όπως η Ιταλική κυβέρνηση. Κάποιοι προβλέπουν ρυθμούς ανάπτυξης πιο μικρούς από αυτούς που προβλέπουμε εμείς. Αυτό δικαιολογεί ένα διάλογο, να γίνονται σεβαστές απόψεις. Ελπίζουμε να δώσει καρπούς ο διάλογος και ο καθένας θα καταλάβει τη θέση του αλλού. Δεν αφισβητούμε την ομιμότητα της κυβερνήσεως της πολιτικές που ακολουθεί. Αλλά εφαρμογή των κοινών κανόνων. Αυτό θέλουμε. Να εφαρμόζονται με ευελιξία, με ευφυΐα αλλά γίνονται σεβαστοί οι κανόνες και να, η ερμηνεία των κανόνων που ισχύουν να είναι η ίδια για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πιέρ Μοσκόβηση, κυρία Ατζέα. Μπορείτε να δείτε και τη πολιτική των ε, προηγούμενων επιτροπών που πραγματικά ε, προέβαλαν πολιτικές λιτότητας. Ενώ τώρα βρίσκουμε μία άλλη οδό. Γκούναρ ε, Χοκμάρκ. Ευχαριστώ. Έχω λοιπόν τις εξής ερωτήσεις. Πρώτον, να πω πως με εκπλήσει πάντα το ότι πρώτα έχετε ένα 100% το οποίο επιτρέπει έτσι δαπάνες λιγότερο σημαντικές. Μετά έχουμε ένα 3% το οποίο προορίζεται για πιο σημαντικές δαπάνες και για τις σημαντικότερες όλων το έλλειμμα ε, μεγαλώνει περισσότερο από όσο επιτρέπεται. Ε, θα μπορούσατε λοιπόν κύριε Πίτροπε, να μου το εξηγήσετε αυτό και να μας πείτε πώς μπορείτε να αντιστρέψετε αυτήν την τάση. Όταν δηλαδή τα, τα, τα κρατημέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν το 100% για να δίνουν προτεραιότητα εκεί που πρέπει. Δεύτερον, εάν η Ιταλία αυξάνει το διαρθρωτικό έλλειμμα και συνεχίσει να το αυξάνει, θα λάβετε μέτρα ή θα βρείτε κάποια δικαιολογία. είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθοριστική σημασία για τα κρατημέλη να γνωρίζουν, διότι έχουμε δει στο παρελθόν με το παλαιό σύμφωνο σταθερότητας ε, πως ε, είχε ορισμένες αδυναμίες, θεωρούταν πολύ ήπιο και νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σέβεται αυτές τις απόψεις και έρχομαι στο επόμενο σημείο που θα ήθελα να τονίσω. Έχουμε μία μοναδική, θα έλεγα, νομισματική πολιτική με μοναδικά ελλείμματα. Τι θα λέγατε λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας για το έλλειμμα και ποια είναι η άποψή σας για το ότι αρκετά κράτη-μέλη δεν συμμορφώνονται με τους ε, απότερους στόχους, συμμορφώνονται με τους ε, ενδιάμεσους στόχους, όμως έχουν ε, τεράστια ελλείμματα. Πώς μπορούμε να επιστρέψουμε σε φυσιολογικά επίπεδα, σε 2,5% επιτόκια. Πώς ε, θα διαμορφωθεί λοιπόν η εικόνα της ε, οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Πρώτα, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δαπάνες, αυτό το 100% συν 3% συν. Όπως είπα και στην αρχή, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, μην το κοιτάξετε παράγραφο-παράγραφο, δείτε το ως σύνολο. Ε, τι επιφέρει μία ισορροπία σε όλον τον κύκλο της οικονομίας. Αυτό θα συμφωνούσατε κι εσείς πως είναι μία λογική προσέγγιση. Έτσι λοιπόν το 3% είναι ένα φράγμα. Υπεραπλουστευμένο βέβαια, αλλά αυτό το 3% είναι ένα όριο, ένας στόχος. Θα έλεγα λοιπόν πως το σκεπτικό πίσω από αυτό είναι ο, ακριβώς αυτή του η θέση στον κύκλο της οικονομίας. Και μετά οι εξελίξεις του λόγου ε, χρέους ΑΕΠ. Ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι αρκετά ε, υψηλότερα από το 60%. Ο στόχος είναι 85%. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη απόκληση ακόμα. Γι' αυτό και οι δημοσιονομικές συστάσεις για την Ευρωζώνη απευθύνονται ακριβώς στα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία έχουν υψηλό ε, λόγο χρέους ΑΕΠ και καλούνται να τον μειώσουν. Αυτά, αυτά αναφέρουν και οι δημοσιονομικές μας συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, αλλά και οι γενικότερες συστάσεις μας ε, για όλη την Ευρωζώνη. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε να κρατήσει για πάντα αυτή η νομισματική πολιτική. Όπως γνωρίζετε, ο πληθωρισμός ε, πέφτει κατά το 2% και εκεί είναι η διαφορά. Αυτό δίνει όθηση στην, ε, και καθορίζει την νομισματική πολιτική και όχι η δημοσιονομική θέση των κρατών μελών. Φυσικά και τα κρατημέλη οφείλουν να προετοιμαστούν για την σταδιακή εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Πολ Τάγκ έχει το λόγο. Δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου όμως. Θα λάβατε μέτρα εάν αυξήσει το διαθροτικό έλλειμμα η Ιταλία γιατί πάντα βλέπουμε πως αυξάνεται, αυξάνεται. Ναι, ναι, ναι, πράγματι, πράγματι, έχετε δίκιο, κάνετε και αυτή την ερώτηση. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει λάβει μέτρα, ήδη έχουν ε, γίνει διαπιστώσεις για σοβαρή μη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει μία διαδικασία ε, υπερβολικού ελλείμματος. Έχει συσταθεί η αντίστοιχη επιτροπή, έχει συζητηθεί στο Eurogroup ε, το έβριμα αυτό και αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε τα επόμενα μέτρα. Βρισκόμαστε σε διάλογο με τις Ιταλικές αρχές και ελπίζουμε να προβούν σε σημαντικές διορθώσεις της δημοσιονομικής τους πορείας. Και κατόπιν θα λάβουμε τα επόμενα μέτρα και θα γίνει τα επόμενα βήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάτι άλλο. Η υπερχείληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται με, την, ε, με τον ε, φορολογικό σχεδιασμό και πώς επηρεάζονται η μία χώρα από την άλλη. Βλέπουμε ας πούμε πώς Υπάρχουν μεγάλε διαφορέ ω προ το κόστο. Η Ιρλανδία έχει 70 δισεκατομμύρια, οι κάτω χώρε 40 δισεκατομμύρια. Αυτό δημιουργεί ανισότητε στου φορολογούμενου. Δεν θα έπρεπε να συμπαριλαμβάνονται και αυτά τα στοιχεία στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Και γιατί δεν υπάρχουν συστάσει αναχώρα ακριβώ για αυτό το θέμα. Δεν γίνεται να υπάρχουν φορολογική παράδειση όπως η Ιρλανδία, η Μάλτα, οι κατοχώρες ε, και να προκαλούν δυσάρεστες επιπτώσεις για τις υπόλοιπες, οι οποίες πρέπει να απομιστούν και το κόστος ε, αυτής της ε, φορολογικής πολιτικής. Έπειτα, αυτές οι πολιτικές ε, θα εξεταστούν από την Επιτροπή. Κύριε Τάγκ, γνωρίζετε πως Ήδη συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για, αυτόν τον, για αυτήν την επιθετική φορολογική πολιτική και φορολογικό σχεδιασμό. Το έχουμε δει, το έχουμε κάνει και στο πλαίσιο των συστάσεων αναχώρα και έχουμε δει, έχουμε διαπιστώσει μάλλον ότι με τεχνικούς όρους δεν υφίσταται φορολογικός παράδεισος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται με ε, τους κανόνες, όλα τα κρατημέλη ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες. Δεν μπορούμε επομένως να ε, πούμε πως έχει διαπιστωθεί ύπαρξη φορολογικών παραδείσεων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς αναφερθήκατε σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες οι οποίες υιοθετούν πρακτικές που θα μπορούσαν να ε, θεωρηθούν επιβλαβείς ή επιθετικές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε στάδιο κατάρτισης μιας έκθεσης που θα προβεί σε, βάθ, σε ανάλυση ε, με μεγάλες λεπτομέρειες αυτών των ε, πρακτικών και φυσικά θα δούμε και η μας τι έχει γίνει για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Νομίζω πως το μήνυμά μας έχει γίνει αντιληπτό και ορισμένα κράτη-μέλη ήδη έχουν επίγνωση του ότι πρέπει να λάβουν μέτρα για να διορθωθεί αυτή η επιθετική φορολογική πολιτική. Να είστε σίγουρος όμως η μάχη, ε, ο πόλεμος δεν τελείωσε. Ευχαριστώ. Τώρα πρέπει να βιαστούμε λίγο, να ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον Στέφαν Γκέρολντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι Επίτροπη. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμεινού, θα, η, δεσμη, δέσμη μέτρων θα έπρεπε να συνεισφέρει στην διασφάλιση της σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από λίγες εβδομάδες ε, αναφέρατε πως ε, η περίπτωση της Ιταλίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις ε, στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης από την Ιταλία. Νομίζω πόσο η επίσης πόσο ο προϋπολογισμός της Ιταλίας δεν είναι ελληματικός ε, τώρα. Υπάρχει αυτή η τάση εδώ και χρόνια. Απλά έχει αλλάξει κατηγορία και αυτό δεν θα επηρεάσει πλέον μόνο τους ε, πολίτες της Ιταλίας αλλά και όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν επίσης πολιτικές λιτότητας που ακολουθούνται εδώ και αρκετά ε, χρόνια σε άλλα κατημέλη. Λένε πως η πολιτική λιτότητα έχει επιβαρύνει την κατάσταση. Αυτό δεν το πιστεύω. Νομίζω πως το ζητούμενο εδώ είναι η εξοικονόμηση πόρων. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Είτε επειδή θέλεις να εξοικονομήσεις πόρους για να κάνεις ένα μεγάλο έργο ή, να, για να, ή επειδή αναγκάζεσαι διότι έχεις άλλα προβλήματα. Στην περίπτωσή μας πρόκειται για την δεύτερη περίπτωση. Βλέπουμε επίσης ότι η λιτότητα και η εξοικονόμηση πόρων ε, δεν είναι ο μπαμπούλας. Ε, δεν φταίει ούτε η καγκελάριος Μέρκελ, ούτε η Λαγκάρτ όταν επιβάλλονται κυρώσεις και πολιτικές λιτότητες σε ορισμένα κράτη-μέλη. Υπάρχουν όμως κάποια λαμπρά παραδείγματα καλών ε, πολιτικών μεταρρυθμίσεων ε, στην Ευρωζώνη, όπου έχουν οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στον ευρωπαϊκό προπολογισμό χώρες της Βαλτικής, για παράδειγμα Σλοβακία. Στην περίπτωση της Ιταλίας πρόκειται για μια διαφορετική περίπτωση. Έχουμε μια κυβέρνηση που αποφάσισε να ασκήσει άλλου είδους πολιτική και αυτό το θεωρούμε λυπηρό η δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έπρεπε να είναι επικεντρωμένη στο πρόβλημα, αλλά στη λύση. Και δεν θα έπρεπε επίσης να εστιάζει σε τίποτα άλλο παρά σε μια βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική. Θεωρώ πως ε, χρειάζεται επίσης ε, να υπάρχουν συνοδευτικά μέτρα που θα στηρίξουν αυτούς τους μηχανισμούς σταθερότητας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση, θα υπάρξει μια ξεκάθαρη απάντηση στις ε, φωνές του λαϊκισμού οι οποίες απαιτούν να ακουστούν και να ακολουθηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο σκέψεις. Μιλήσατε για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ικανότητα μεταρρύθμισης σε ορισμένες χώρες. Τώρα τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν κάτι διαφορετικά. Όμως υπάρχουν, υπάρχει και αυτή η όθηση σε επίπεδο συμβουλίου. Για την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το ΕΚΟΦΗΝ και το Eurogroup και εσείς θέσατε επιτάπητος το θέμα της μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης και μιλήσατε και για αυτή την δημοσιονομική ατζέντα που προώθησε ο Επίτροπος Μοσκοβισή. Μιλήσαμε για την ασφάλεια των καταθέσεων, για, τον, για το backstop, για το μηχανισμό ασφαλείας ε, του Ταμείου Εξυγίανσης και ένα γενικότερο όριο διαφορετικά δεν είναι backstop. Επίσης μιλήσατε για την προστασία των επενδύσεων, για τις ε, αντικυκλικές τάσεις. Μιλήσαμε και για το, τους ψηφιακούς φόρους, τον ψηφιακό φόρο, την παγιοποίηση των λογαριασμών. Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι υπάρχει τάση μεταρρύθμισης και η Επιτροπή δεν μπορεί να περιμένει και να πιέζει το Συμβούλιο τους υπόλοιπους μήνες για να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Το δεύτερο έχει να κάνει με την έλλειψη ικανοποίησης πολλών κρατών μελών. Είπατε δηλαδή ότι η Ευρωζώνη ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία. Ο δείκτης ανεργίας κατεβαίνει, όμως στη Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία βλέπουμε ότι αυτή η βελτίωση, παρά τη βελτίωση αυτή, ε, δεν μπορούμε να περάσουμε αυτή την ανάπτυξη στους πολίτες. Και ποια είναι τα μέτρα που προτείνει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση στα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα στους πολίτες. Ντανούτα Χούμπνερ. Ευχαριστώ. Για μένα η Ιταλική περίπτωση δείχνει τη σημασία της εθνικής κυριαρχίας, αν θυμάμαι καλά, μετά την έκθεση των πέντε προέδρων το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου άλλαξε κάπως για περισσότερες συζητήσεις στα Εθνικά Κοινοβούλια και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να βελτιώσετε αυτό τον διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Κοινοβουλίων για τους δημοσιονομικούς κανόνες. Σε σχέση τώρα με την αυτονομία των δημοσιονομικών ευρωπαϊκών φορέων, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο είναι πραγματικά ανεξάρτητοι αυτοί οι εθνικοί οργανισμοί ε, δημοσιονομικής αποτίμησης. Θεωρείτε ότι το σύστημα έχει βελτιωθεί χάρη στους, ε, στους οργανισμούς αυτούς, στα διοικητικά συμβούλια και υπάρχει συνεργασία μεταξύ εθνικών θεσμικών οργάνων και ευρωπαϊκών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ερωτήσεις. Θα αναφερθώ σε κάποιες στοιχείες εγώ και κάποιες άλλες θα αφήσω στον Πιέρ. Σχετικά με τη γενική συζήτηση. Δηλαδή, ποια γενική δημοσιονομική πολιτική είναι η ενδεδειγμένη στις οικονομικές περιστάσεις και το πλαίσιο αυτό. Επί του παρόντος, έχουμε μια ουδέτερη δημοσιονομική τοποθέτηση του χρόνου, βλέποντας το συνδυασμό δημοσιονομικών σχεδίων προπολογισμού των κρατών μελών της Ευρωζώνης θα δούμε μία επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Από την πλευρά μας συστήνουμε η, κανή, καλή αυτή οικονομική περίοδος να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσουμε ε, δημοσιονομικά μέσα απορρόφηση των κραδασμών και αυτό θα προτείνουμε και στις εκθέσεις αναχώρα στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι κατεπήγον αυτό με υψηλά ποσοστά χρέους προς ΑΕΠ. Και επανειλημμένα το τονίζουμε αυτό. Για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Αναφερθήκατε στη Σλοβακία και τις χώρες της Βαλτικής. Λειτουργούν οι μεταρρυθμίσεις και οι χώρες που εφαρμόζουν φιλόδοξες διαθροτικές μεταρρυθμίσεις είναι ανάμεσα σε αυτές που αυξάνονται με πολύ ψηλού ρυθμούς. Θα μπορούσα να προσθέσω την Ιρλανδία και την Ισπανία και την Πορτογαλία. Βλέπουμε ότι χώρες που εφάρμοσαν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει βελτιώνουν και τους δείκτες ανάπτυξής τους. Κάποιες άλλες ερωτήσεις που ετέθησαν και αφορούσαν την εμβάθυνση των αποτελέσματα του Eurogroup και της δεν θέλουμε να προδικάσουμε τις αυριανές συζητήσεις επί του θέματος. Πιο συγκεκριμένα θέματα, όπως για το Ταμείο Αξιολόγησης των Σημείων Υποστήριξης και για το μηχανισμό σταθερότητας βρήκαμε μεγαλύτερη πρόοδο, αλλά όσον αφορά τα δημοσιονομικά μέσα, το πρόγραμμα υποστήριξης των Ταμείων και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Σταθεροποίησης είδαμε λιγότερη πρόοδο αλλά έχουμε κάνει προτάσεις και θα τις συζητήσουμε και θα διευκολύνουμε τη συζήτηση. Το ίδιο και γι' αυτό τις τρα, τα, τραπεζικές εγγυήσεις για τα κρατικά ομόλογα έχουμε προτάσει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν υπάρχει πρόοδος στο Συμβούλιο και δεν έχει ψηφιστεί και έκθεση του Κοινοβουλίου, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου. Σε κάποια φάση θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στη συζήτηση για τους δημοσιονομικούς κανόνες. Κατά πόσο τους ενστερνίζονται οι διάφορες χώρες και εθνικοί αρμόδιοι φορείς και ευρωπαϊκοί φορείς. Βλέπουμε να υπάρχουν αποτελέσματα. Υπάρχει ανεξάρτητη τοποθέτηση επιδημοσιονομικών προγραμμάτων των κυβερνήσεων και ανεξάρτητη άποψη όσον αφορά την κατάσταση στην Ευρωζώνη. Είναι τα πρώτα βήματα που είδαμε από το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και από τους εθνικούς δημοσιονομικούς φορείς και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το πλαίσιο είναι χρήσιμο. Είναι νεότευκτο το πλαίσιο, δεν μπορούμε να συναγάγουμε τελικά συμπαράσματα σε αυτή τη φάση. Τα πρώτα βήματα είναι ενθαρρυντικά και θα πρέπει να συνεχίσουμε την ενίσχυση των θεσμών αυτών και να ισχυροποιήσουμε τη φωνή τους στις διάφορες συζητήσεις για τα δημοσιονομικά. Λίγα να προσθέσω, λέει ο κ. Μοσχοβησί, έχω. Θα επικεντρωθώ επί τη τελευταία πτυχή. Απαντώντας τον κύριο Φερνάντες. Γιώνας. Το Eurogroup τη περασμένη Εβδομάδα ήταν δύσκολο. Κράτησαν πολλοί συζητήσει, πάρα πολύ. Και καταλήξαμε σε κάποιες προτάσεις που έχουν τρία θετικά στοιχεία και έχουν και όρια βέβαια. Τα, τα θετικά στοιχεία. Οι υπουργοί της Ευρωζώνης έθεσαν πρόγραμμα εργασιών φιλόδοξο το Σεπτέμβριο. Και συστημικά το υλοποίησαν, συστηματικά το υλοποίησαν. Και πρώτε αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων που συνεδριάσουν την πέμπτη, τη μορφή ευρωζώνη μια δέσμη μέτρων. Οπότε έχει εκτελεστεί η αποστολή του Eurogroup. Άλλες, άλλα δύο σημεία στα οποία προοδεύσαμε. Το πρώτο αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητος. Η Ρίστον Παρόδο ότι ήταν δύσκολη η συζήτηση, κράτησε πολύ, δεν ήταν και απλή. Ενεκρίθη αυτός ο μηχανισμός από το Eurogroup και επιτρέπει ενίσχυση του ρόλου σύμφωνα με την πρότασή μας. Θέλαμε για το ενιαίο μηχανισμό ε, εξυγίανσης να έχει κάποια υποστήριξη. Backstop. Ποιο ήταν το όριο το έντις, την ασφάλεια των καταθέσεων. Ήταν ο τρίτος ε, πυλώνας τραπεζικής ενώσεως ε, αρχικά. Ήταν πρωτοβουλία του Βάλης Ντομπρόφσκης. Παραμένει επιτάπητος η πρόταση. Αυτός ο τρίτος πυλώνας θεωρούμε ότι είναι αναγκαίος. Γι' αυτό πολιτικός προβληματισμός και τεχνικές συζητήσεις είναι καλός ιονός. Θα θέλαμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα πιο μακριά και κάποια προκαταλήψεις μας σταματήσουν και κάποια μπλοκαρίσματα. Πολιτικός στόχος σημαντικός ε, τα οικονομικά της Ευρωζώνης. Η κυρία Περές και ο κ. Μπέγκε το επεξεργάζονται. Από την αρχή της θητείας το εξετάζαμε το θέμα. Ακόμα πολλά απομένουν να γίνουν για τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Υπάρχει η πτυχή της ανταγωνιστικότητας και για το Ταμείο Σταθεροποίησεως. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία γι' αυτό. Αυτό πρέπει να ξαναπροωθηθεί. Χωρίς προπολογισμό η Ευρωζώνη είναι δύσκολο να θεωρηθεί ότι έχει πραγματοποιήσει μεγάλη μεταρρύθμιση. Το μπαλάκι είναι στα χέρια των αρχηγών κρατών κυβερνήσεων και ελπίζουμε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Όσο μας αφορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τέλος της θητείας θα εξακολουθεί να παίζει το ρόλο της, να προωθεί τις προτάσεις της. Καμία πρότασή μας δεν έχει αποσυρθεί. Όλες είναι επιτάπητος, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου σταθεροποίησης. Δεν θεωρούμε ότι έχει παραμεριστεί, θα σφάλμα. Χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τους ασύμετρους κλειδονισμούς της Ευρωζώνης. Διαφορετικά δεν θα είχε νόημα και ένας προπολογισμό της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει και ο Σύντομα τελικά σχόλια από τον εισηγητή μας, τον Τόμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα πάρα πολλά για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, και την περίπτωση της Ιταλίας. Όμως ε, φάνηκε κάτι ιδιαίτερο από αυτήν την ε, συζήτηση. Πόσο περίπλοκη είναι αυτή η κανόνες και ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης οφείλει να δώσει ε, διαφάνεια, να κατευθύνει. Όμως ε, βλέπουμε πως ε, συμβαίνει το αντίθετο. Δημιουργούνται εμπόδια, ασάφειες. Στην έκθεσή μου προσπάθησα να επικεντρωθώ στη σημασία που έχουν τα ανοιχτά καθαρά γη δημόσια οικονομικά. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να υπάρχει ένα απόθεμα αντιμετώπισης του κινδύνου και φυσικά να υπάρχουν σαφείς ε, κανόνες, οι οποίες όμως δεν θα είναι πολύ ε, περίπλοκοι. περίπλοκη. Τέλος, ε, αναφέρομαι στην ευελιξία που πρέπει να υπάρχει στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να μπορεί να ασκείται υγιής δημοσιονομική πολιτική και να γίνονται παραγωγικές επενδύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως ε, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και είναι, πιστεύω πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε το βήμα που μας δίνει αυτή η Επιτροπή για να συζητούμε όχι μόνο γενικότερα οικονομικά ζητήματα αλλά και ε, έκτακτες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα την περίπτωση της Ιταλίας. Να ευχαριστήσω ξανά τους Επιτρόπους κ. Ντομπρόφσκης και Μοσκοβισή και εύχομαι να έχουμε θετικές εξελίξεις όχι μόνο στην ε, περίπτωση της Ιταλίας, αλλά γενικότερα όσο προς την ε, εφαρμογή ε, της δημοσιονομικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αύριο θα γίνει μια πολύ σημαντική συζήτηση στην Ολομέλεια για την μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Θα θέλατε όμως, κυρία Μπαρέση, να, να σχολιάσετε αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας. Οι αντιπρόεδροι εδώ έκαναν μία τριπλή παρουσίαση. Ε, την κατάσταση στην Ιταλία, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη. Θα έχουμε όμως και μία άλλη συζήτηση στην έκθεση του συναδέλφου από το ΕΛΚ γιατί οι άλλοι σκιώδεις δεν ε, πήραν το λόγο. Ναι. Θα το εξετάσουμε προσεκτικά. Έχει ήδη προγραμματιστεί η εξέταση ανθρωπολογιών τον Φεβρουάριο. Δεν χρειάζεται να παρουσιαστούν αυτά. Ναι, κατάλαβα, ήσασταν σαφείς. Η συζήτηση για την έκθεση ήταν μια συγχώνευση, μια σύμφυση πολλών θεμάτων, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Φυσικά και θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης τον Ιανουάριο. Σας ευχαριστώ. Έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό, κύριε Περέιρα. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, τον Ιανουάριο θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι. Οι τροπολογίες πρέπει να παρουσιαστούν μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Και σύμφωνα με την συνήθεια διαδικασία, πρώτα γίνεται μία ανταλλαγή απόψεων και έπειτα η παρουσίαση των τροπολογιών. Yes, thank you. No, I think... Σας ευχαριστώ. Όντως, πολύ εύστοχο το σχολείο σας γιατί στις 25 Φεβρουαρίου προβλέπεται η εξέταση των τροπολογιών. Και φυσικά πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο, να δούμε αν έχουμε χρόνο, διότι αν εξετάσουμε τις τροπολογίες τέλος Φεβρουαρίου, όπως αναγράφεται εδώ στο πρόγραμμα, νομίζω πως χρειάζονται δύο μήνες ή και παραπάνω από την ημερομηνία που κατατίθενται οι τροπολογίες και την ημερομηνία που εξετάζονται. Τόμ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το αρχικό σας σχόλιο, όταν είπατε δηλαδή ότι θα ενώσετε πολλά θέματα για να γίνει συζήτηση, είναι η εφορμή που παίρνω το λόγο, θα μπορούσαμε λοιπόν βέβαια να το κάνουμε αυτό, όμως δεν θέλω να τραβήξει η διαδικασία παραπάνω από όσο χρειάζεται. Έπειτα, καλώ τους και όδους συζητητές να μου στείλουν σχόλια ή και διμερώς αν θέλουν να το συζητήσουμε, να αρχίσουμε να δουλεύουμε το φάκελο αυτό για να μην χρονοτριβούμε. Όχι, δεν χρονοτριβούμε. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου. Δεν αλλάζει κάτι γι' αυτό στην ημερομηνία της ψηφοφορίας. Θέλουμε να σας δώσουμε την ικανότητα, τη δυνατότητα να συζητήσετε με τον κύριο Πίτροπο και φυσικά να έχετε το χρόνο να συζητήσετε την έκθεσή σας, κάτι που δεν ε, ήταν δυνατόν σήμερα. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε ό,τι καλύτερο δεδομένης της κατάστασης. Ευχαριστούμε πολύ τους Επιτρόπους κ. Ντομπρόφσκης και Μοσκοβισή. Διακόπτουμε για ένα λεπτό και μετά περνάμε στις ψηφοφορίες. Μόνο για να πάρετε τους καταλόγους ψηφοφορίας. Συνάδελφοι, Okay. Λοιπόν, ας κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Τεστ, ψηφίζουμε. Άρχεται η δοκιμαστική ψηφοφορία. Πέρας. Λοιπόν, ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης για τη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά, συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ κατά απόφυγες εγκρίνεται, τροπολογία 82 υπέρ κατά απόχες, ελέγχουμε την 82. Πέρας. Απορρίπτεται. 26 ψήφοι κατά. Συμβαστική αλφά-αλφα Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 87. Υπέρ κατά, αποχές Το 88 υπέρ, κατά, αποχές Το 89 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτω. 20 υπέρ. Α, από την 89 θέλετε να την ελέγξουμε. Πολύ ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, είστε υπέρ. Θα το εγκρίνετε τότε. Πέρας. Εγκρίνεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές όχι θέλετε έλεγχο 104 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά έλεγχο στην 29 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1 υπέρ. Καλύπτεται λέτε. Ναι, ναι, ναι, είναι συμβατή. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Νομίζω πως κάτι έχει ο κατάλογός μας, πάρω έναν άλλο καλύτερα, τα βλέπω καλύτερα. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά εγκρίνεται, 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά εγκρίνεται κατά 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 8 εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ έλεγχο στην 66. Vote is closed. Πέρας, εγκρίνεται. 26 υπέρ, 21 κατά, 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ Απορρίπτε. Συμβαστική DA ε, υπέρ κατά εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές, έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Πέρας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική, όχι, τροπολογία 71, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική DB, υπέρ, κατά, αποχές, απο... εγκρίνεται. 72, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 73, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 απορρίπτεται 76 υπέρ κατά απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά έλεγχος 15 Πέρας εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 41 ψήφοι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 Αρχικό κείμενο υπέρ κατά εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ κατά έλεγχος της τροπολογίας 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος της τροπολογίας 7. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά έλεγχος πέρας. 38 ψήφι υπέρ εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο, ψηφίζουμε το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 48 υπέρ, 0 κατά 0 αποχές, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ψηφίζουμε για τα benchmark την Πέμπτη. Γίνεται κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και συζήτηση και ψηφοφορία για το benchmark την Πέμπτη. Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα σας.